Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, λέει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Και στα αγγλικά τώρα, παρακαλώ καθίστε. Σε μισό λεπτό αρχίζουμε. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego przerwanego w dniu 8 lipca 2010 roku. Συνεχίζουμε τις εργασίες, της ολομιλίες της 8 Ιουλίου. Όλοι ορίσατε. Καλό χειμώνα, ελπίζω ότι ξεκουραστήκατε στις διακοπές, γιατί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και τώρα μερικά ενημερωτικά. Σας επισημαίνω ότι η κυρία Σακίνη Ασιάδη, η οποία καταδικάστηκε εις θάνατο στο Ιράν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, ε, πέτυχε την ακύρωση της απόφασης από το ανώτατο δικαστήριο. Υπέστη